σύνορα με την πλήρη απομόνωση. Και ε, έτσι καταδιώκουν ανθρώπους ε, και τους στέλνουν στα χέρια των διακινητών. Η, τα, η, η απόρρια αυτής της πολιτικής φαίνεται στη Λιβύη τώρα. δεν φτάνει ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν αναλαμβάνουν τις χριστιανικές τους ε, ευθύνες, αλλά αν ε, ακολουθούσαμε τους ε, συντηρητικούς θα έπρεπε να ε, αναθέσουν τις επιστροφές σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μεταθέτει δηλαδή ίδιες ευθύνες σε άλλους. Αυτό το απορρίψαμε με επιτυχία. Το Συμβούλιο που λάμπει σήμερα δια της απουσίας του πότε θα ε, ολοκληρώσει ένα πακέτο για το ε, άσυλο που θα είναι ισορροπημένο. Πότε θα υπάρξουν ενιαίοι κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο βιώσιμο και μακροπρόθεσμο τις προκλήσεις στα σύνορα και θα ε, ανταποκριθούμε και όπως πρέπει στις κοινέ μας αξίες. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Σόιντροβα. Οπωσδήποτε όχι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ε, Μπέρντ Κέλμελε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση η Frontex και προσωπικό περισσότερο χρειάζεται. Είναι σωστό το μέτρο. Παράλληλα, ε, οι 10.000 ε, δημιουργούν ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα της Ένωσης δεν θα τα λύσουμε ε, ζητώντας μόνο περισσότερα χρήματα. Αυτό που χρειάζεται για τη μετανάστευση είναι μία ρύθμιση νομοθετική ευρεία που θα δώσει ε, τη δυνατότητα ανάληψης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο έλεγχο στα σύνορα, πρέπει να μπορούμε να αποφασίζουμε ποιος μπορεί να μπαίνει και ποιος δεν μπορεί να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εδώ έχουμε μια πλειοψηφία που αναζητεί απλές λύσεις και νομίζει ότι θα καλύψει τα προβλήματα με λεφτά. Ενώ τα προβλήματα στην πραγματικότητα επιδεινώνονται και οι νέοι δεν θα είναι έτοιμοι όταν θα ξεσπάσει νέα κρίση και αυτό σίγουρα δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Αν θέλουμε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στους πολίτες πρέπει τη βούληση των πολιτών να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας στα σοβαρά και χρειάζεται να γίνει κάποια στιγμή μια σωστή συζήτηση για αυτό το θέμα. Η κυρία Βίξτρομ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο Ρομπέρτα Μέτσολα για την πολύ καλή δουλειά τη. Σα ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ετών. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την πολύ καλή αυτή πρόταση. Όταν πετάω στην Ευρώπη, εγώ δεν βλέπω σύνορα. Αυτό το είχε πει ο πρώτο πρόεδρο τη ελεύθερη Τσεχοσλοβακία, ο Βάκλαβ Χάβελ η μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής ένταξης, η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, βασίζεται στο να έχουμε ισχυρά εξωτερικά σύνορα. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη οχυρό. Δεν θέλουμε να διώξουμε ανθρώπους. Θέλουμε να ελέγχουμε τις ροές των ανθρώπων που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται ένα σωστός έλεγχος ασφαλείας, υπάρχει μια διέλευση συντεταγμένη για όλους όσους έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας ε, ε, ε, διεθνή προστασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών, παράνομων ουσιών που δεν θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση που εγκρίνουμε σήμερα δεν πάει προς ένα πλήρες ομοσπονδιακό σύστημα. Για μένα αυτό είναι ο σωστός δρόμος, αλλά έχουμε γίνεται ένα πρώτο βήμα από τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι εγώ είμαι δέκα χρόνια εδώ. Είναι από τι τελευταίε μου ομιλίε ε, στην Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου, όλου όσου με του οποίου συνεργάστηκα. Ε, όταν τελειώνει η πολιτική, η φιλία μένει. Και είναι μια ευκαιρία και μια νέα αρχή. Ευχαριστώ. You are an optimist. Sometimes politics. Είστε αισιόδοξοι. Καμιά φορά η, η πολιτική καταστρέφει φιλίες, τέλος πάντων. Ελπίζω να ισχύσει αυτό που λέτε στην προηγουμένη περίπτωση. Η κυρία Φορέντζα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 1.311 θάνατοι μόνο και μόνο το 2018. Αυτό είναι ο απολογισμός των θανάτων στη Μεσόγειο. Και εμείς συνεχίζουμε και συζητάμε εδώ πέρα για σύνορα και για ενίσχυση της πολιτικής επιστροφών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Καταρχάς, θα πρέπει να κηρύξει ως μη ασφαλής τους λιμένες της Λιβύης. Το έχει κάνει αυτό επίσημη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχουν κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούν ότι είναι ασφαλεί οι επιστροφέ στη Λιβύη και στι χώρε αυτέ συγκαταλέγεται και η Ιταλία. Αν πραγματικά θέλουμε να μας θυμόμαστε, να μας θυμάται ο κόσμος ως αυτοί που αύξαν τους θανάτους στην Μεσόγειο, τότε δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό. Το αντίθετο όμως θα έπρεπε να ελπίζουμε. Σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραπέμπουμε στις λιβικές αρχές την όλη αρμοδιότητα και ευθύνη της έρευνας και της διάσωσης. Καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία με την αστευτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ακολουθούμε την πολιτική του Σαλβίνη, πρέπει να είμαστε μια πολιτισμένη Ήπειρο. Η κυρία Βαλέρο έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για του πρόσφυγες, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που φεύγουν από τι χώρε του εξαιτία ένοπλων συγκρούσεων και από ό,τι φαίνεται η τάση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Θα έχουμε όλο και μεγαλύτερα μεταστευτικά κύματα εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε εκατομμύρια κλιματικών λεγόμενων προσφύγων και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τους 600.000 ε, πολίτες οι οποίοι θα πληγούν λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσας σε διάφορες χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να έρθουν προς την Ευρώπη, όχι όλοι βέβαια, αλλά εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν προς, την Ευρώπη. Επενδύουμε αυτή τη στιγμή τεράστια ποσά προκειμένου να τους απομακρύνουμε, προκειμένου να τους κρατήσουμε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έπρεπε να τα δίνουμε για την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών, αλλά περισσότερο για τη μείωση τη φτώχεια και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσή του. Ο κύριο Κορά έχει το λόγο τώρα για μισή λεπτό. Α το πούμε ξεκάθαρα, αγαπητοί συνάδελφοι, απέτυχε η μεταρρύθμιση του κοινού συστήματο ασύλου. Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια τίποτα δεν έγινε προκειμένου να τροποποιηθεί η Συμφωνία του Δουβλίνου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι βυθίζεται σε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο η Λιβύη και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ζωές από τη Λιβύη. Νομίζω ότι η Frontex αυτή τη στιγμή είναι το μόνο εργαλείο το οποίο έχει απομείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικεύει το, πρόβλημα αυτό, δίνει χρήματα σε τρίτες χώρε για να κάνουν αυτέ τη βρώμικη δουλειά. Και από την άλλη η μεταρρύθμιση του Frontex συνάδει ουσιαστικά με την πολιτική αυτή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ελπίζουμε μέσω της μεταρρύθμισης αυτής, ελπίζουν ορισμένοι τουλάχιστον, να κερδίσουν περισσότερες ψήφους στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Ανταυτού όμως θα έπρεπε να είχαμε περισσότερη ευρωπαϊκή ελληνική, την οποία όμως δεν θέλουν καν να ακούσουν, ούτε καν ως ιδέα, ως έννοια, ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ενισχυθούν περισσότερο οι χώρε εκείνε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίε καλούνται να διαχειριστούν τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω επίσης ότι ε, στις ε, χώρες αυτές θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν ακόμα και εσωτερικούς ελέγχους, τη στιγμή που τους ελέγχους αυτούς δεν μπορεί να κάνει ο οργανισμός, ο Frontex. Κανονικά η αρχή τη αλληλεγγύη υποτίθεται ότι προβλέπεται από τι συνθήκε, αλλά στην πράξη δεν ισχύει, δεν λαμβάνει χώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Επιτήδιος. Παρά το γεγονό ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη πω το Frontex είναι το πλέον ανεπιτυχέ πείραμα για να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να τον αναβαθμίσει και να τον μετατρέψει σε οργανισμό Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή. Ε, το αυξάνει την επιχειρησιακή δύναμη σε δέκα χιλιάδε άτομα και σε περιόδους αγρίας λιτότητας φορολογεί τους ευρωπαίους πολίτες και σπαταλά τα χρήματά τους για να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό άρα και άχρηστο οργανισμό. η αιμονή όμως και η σκοπιμότητα να αφαιρεθούν από τα εθνικά κράτη αρμοδιότητες ζωτικές για την επιβίωσή τους όπως είναι η ασφάλεια των συνόρων οδηγεί την ευρωπαϊκή ένωση να λάβει αποφάσεις που αντίκειται στην κοινή λογική διότι ποιο λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο θα διαφωνήσει με την άποψη ότι η καλύτερη προστασία των συνόρων ενό κράτου επιτυγχάνεται εάν η αποστολή αυτή δοθεί στι ένοπλε δυνάμει και τα σώματα ασφαλεία του κράτου αυτού. η ορθότητα αυτή τη απόψεω έχει αποδειχθεί στην πράξη διότι όλα τα κράτη τα περισσότερα κράτη τη ευρωπαϊκή ενώσεω κλείνουν τα σύνορά του για να αντιμετωπίσουν τα ανεξέλεγκτα κύματα των λαθρομεταναστών και έτσι μεταφέρουν το πρόβλημα στα κράτη εισόδου όπω είναι η ελλάδα η οποία εάν δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει μόνη της να προστατεύσει τα σύνορά της ουδής μαθητευόμενος μάγος της ευρώπης θα τη βοηθήσει υπό οποιαδήποτε μορφή και όνομα και αν εμφανιστεί αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διάς Δεμέρα τώρα έχει το λόγο για μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, θέλω να συγχαρώ τη Ρομπέρτα για την καλή δουλειά της. Υπενθυμίζω όμως ότι η διαχείριση Τη μετανάστευση με αποτελεσματικότητα και με ένα υψηλό επίπεδο ασφάλεια στο ιστορικό τη Ένωση, Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίω να διαφυλάξουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η δημιουργία ενό σώματο 10.000 ανθρώπων, η υποστήριξη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι επιστροφές ή η εντετικοποίηση τη συνεργασία με τρίτες χώρε είναι πολύ σημαντικά επιχειρησιακά στοιχεία για να εγγυηθούν μια συνεχή υποστήριξη και για τις χώρες προορισμού και για τις χώρες προέλευσης και για τις χώρες transit. Από κοινού με τη Europol αυτή η νέα υπηρεσία θα είναι η λιδία λίθος που θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα χώρο ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια στην Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε το έργο μα για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερε επιχειρησιακέ, να δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερε επιχειρησιακέ και δημοσιονομικέ δυνατότητε σε αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει βεβαίω και μια δικλίδα ασφαλεία. διότι αυτή, αυτό το σώμα υπόκειται στο δίκαιο της θάλασσας, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαγιών έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σίγουρα χρειάζεται καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης αυτό είναι σημαντικό για την καλύτερη λειτουργία του χώρου Σέγγεν, για την ε, ρύθμιση της μετανάστευσης. Χρειάζονται συμφωνίες ε, για την ε, επέκταση και ενίσχυση του Frontex. Θα ψηφίσω υπέρ. Είναι σημαντικό να έχουμε την αύξηση αυτή στις 10.000 μέχρι το 2027. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την βασική ευθύνη για τη διαχείριση των συνόρων τους και θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατέψουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που θα επιστραφούν από τη Frontex στις τρίτες χώρες. Η συνεργασία με τρίτες χώρες ε, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νέων συμφωνιών που θα λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, προσοχή, οι νέοι κανόνε για τα εξωτερικά σύνορα δεν θα πρέπει να ισχύουν χωρί να προσαρμοστούν και για τον ε, ευρωπαϊκό εξωτερικό χώρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαμπάσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σαφώ θα πρέπει όλα αυτά τα χρήματα να δοθούν στο νέο αυτό οργανισμό. Τα εξωτερικά σύνορα είναι θεμελιώδους σημασίας, προκειμένου πραγματικά να έχουμε ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χαιρετίζω την διευρυμένη αυτή αρμοδιότητα που δίνεται στο νέο αυτό Frontex, και είμαι σαφώ υπέρ τη θέσπιση του μόνιμου αυτού σώματο με επιχειρησιακή δύναμη 10.000 ατόμων. Το έχω πει πολλάκι στο παρελθόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού για να σταματήσουμε την έλευση των παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικοί μετανάστε, οι οποίοι δεν δέχονται τι αξίε μα και τον τρόπο ζωή μα, δεν έχουν καμία θέση στι χώρε μα ούτε βέβαια και οι τρομοκράτε, ε, οι οποίοι χρησιμοποιούν πολλέ φορέ τις οδού μετανάστευση. Σα ευχαριστούμε. Ουρτασούν παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η θητεία θα περάσει στην ιστορία για την τροπή των 18.000 νεκρών στη Μεσόγειο σύμφωνα με τη Διεθνή ε, Οργανισμό Μεταναστών και το τελειώνουμε τη θητεία με το χειρότερο τρόπο με, τον, με την μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, του κανονισμού του ασύλου που έχουν μπλοκαριστεί και έχουμε τώρα αυτόν τον νέο κανονισμό για μια ακτοφυλακή στην οριοφυλακή με δισεκατομμύρια που διατίθενται χωρί να υπάρχει ένα μηχανισμό που να διαφυλάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρί μια σαφή εντολή για την διάσωση στη Μεσόγειο όπω έχει ζητήσει αυτό το κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευσή της και στην πραγματική εντολή της το έχουμε ζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν οι κυβερνήσει τελικά ποινικοποιούν τη ΜΚΟ όπω το Open Arms που δεν μπόρεσε, μπόρεσε να ε, φτάσει να, να, να πιάσει λιμάνι στη Βαρκελόνη ε, ποινικοποιούμε λοιπόν τη ΜΚΟ ε, και δεν γίνεται αναφορά σε μια δημόσια προσπάθεια διάσωσης. Είναι πραγματικά μια ντροπή. Στην νέα θητεία θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάλ έχει, δύο, έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η Frontex τη θεωρία ε, θα μπορούσε να προστατεύσει τα σύνορα της Ένωσης Όμω είναι ευθύνη των κρατών μελών κυρίω αυτό. Η ενίσχυση λοιπόν της, ε, των αρμοδιοτήτων τη Frontex ε, είναι κάτι που θα μπορούσε να διακυβεύσει την ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν πρέπει να παρεμποδιστούν τα κράτη-μέλη από το να προστατεύσουν τα σύνορά του. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν συνεργασία. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό στην πράξη. Ανησυχούμε, διότι η συμφωνία που επετεύχθη δεν επιτρέπει στην Frontex να έχει την υποστήριξη των αρχών ε, σε τρίτες χώρες όπως τη Μακεδονία και δεν θα μπορεί να βοηθήσει για την επιστροφή των πάνω μεταναστών. Εμείς θα πάντα να υπάρξει μια ενίσχυση ε, των συνόρων και έχουν καταφέρει εμεί να προστατεύσουμε τα σύνορά μα χωρί την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Η Ουγγαρία όμω δεν είδε ποτέ λεφτά για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Γκυλιόμ. σω να ήταν τελικά απαραίτητο να ενισχυθεί η υπηρεσία Frontex, διότι τα κοινά μα σύνορα πρέπει να τύχουν διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή τη μεταρρύθμιση ε, τη Ευρωπαϊκή, Συνοριοφυλακή, που πρέπει να συνοδεύεται όμω από το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων όσων ελέγχονται στα σύνορα τα εξωτερικά τη Ένωση. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ και σε δύο παράπονα που έχω στο τέλο τη θητεία αυτή. Ε, λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε μία ε, αποστολή διάσωση στη γη πάνω από 1.800 ε, άνθρωποι πέθαναν το 2018. Άνθρωποι κινδυνεύει ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί με τέτοια υπηρεσία να το κάνει αυτό. Ε, εδώ και 6 μήνες οι ΜΚΟ το κάνουν αυτό ε, στην θάλασσα. Ε, κλείνουν τα σύνορα, τα κράτη-μέλη. παρόλα αυτά συνεχίζουν οι μετανάστε να προσπαθούν να περάσουν και βεβαίω υπάρχει δεύτερη μεταρρύθμιση της Frontex, ε, να υπάρχει καμία μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά το καθεστώς ασύλου. Και γι' αυτό λυπάμαι και φταίνουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό που μπλοκάρουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, ενώ το Κοινοβούλιο έχει θέσει τη θέση του επιτάπητο εδώ και δύο χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Τόμα, έτσι και ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Frontex πρέπει να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αλλά είναι λάθος η κατεύθυνση που του δίνουμε του οργανισμού αντί να εξειδικεύεται σε επίγουσες καταστάσεις ε, και γρήγορη αντίδραση, δημιουργούμε γραφειοκρατικές υπηρεσίες τώρα. Είναι αμφισβητούμενο το πόσο θα αποδώσουν. Πρέπει να λύσουμε άμεσα τα προβλήματα. Η Frontex δεν μπορεί να ε, συμμετέχει σε επιχειρήσεις από τρίτες σε τρίτες χώρες. Δεν θα μπορεί να επιστρέψει ε, από τις, βόρειες Ευρω... Ε, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις χώρες από όπου προέρχονται. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να αντιμετωπίζουμε το οργανωμένο ε, έγκλημα και την παράτυπη μετανάστευση ε, στο κατόφλι των χωρών μας, ενώ θα έπρεπε να γίνεται αυτό όσο γίνεται πιο μακριά. Σας ευχαριστούμε κύριο Ρανχέλ για μισή λεπτό παρακαλώ. Πουσιάζει όμως. Η κυρία Κιέγγε για ένα λεπτό τότε παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προώθησε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού που θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοροφυλακή και Ακτοφυλακή. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τι εσωτερικέ διχόνοιε, διαπραγματευτήκαμε και καταλήξαμε τελικά σε ένα κείμενο το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξο, αλλά σίγουρα θα συμβάλλει το να παγιώσουμε έναν από τους τέσσερις πυλώνες που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και αναφέρομαι βέβαια στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια στο πλαίσιο του πυλώνα αυτού καλεί την Ευρώπη να ενισχύσει τη δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Θα πρέπει προφανώ να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επομένως, η υποστήριξη της μεταρρύθμισης αυτής θα επιτύχει μόνο αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά και αν εξασφαλίσουμε επίσης τη δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και να κάνω μια έκκληση στο τέλος της θητείας αυτής. Σας παρακαλώ πολύ, εκινήστε εκ νέου την επιχείρηση Σοφία και δώστε τις μεγαλύτερες δυνατότητε έρευνας και διάσωσης. Ο κύριος Ράντεφ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησα την εντολή μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την εποχή εκείνη η όλη ιδέα θέσπιση ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνορεφυλακή και Εκτοφυλακή ήταν ένα πολύ ασαφέ και θεωρητικό σχέδιο. Θεωρούσαμε ότι θα έβλεπε το φω τη ημέρα το νωρίτερο το 2030. Είμαστε όμω πάρα πολύ αφελεί τότε, γιατί μέσα σε ένα χρόνο είδαμε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστε και πρόσφυγε να καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασχίζοντα τα εξωτερικά μα ε, σύνορα και οι τότε συνοριοφύλακες δεν ήταν σε θέση να διχειριστούν ένα τόσο ακραίο φαινόμενο. Έπρεπε λοιπόν επιγόντω να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μα σύνορα και συνειδητοποίησαμε ότι ο χώρο Σέγγεν είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Συνειδητοποίησαμε τότε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των εξωτερικών τη σύνορων καταρχά και τέσσερα χρόνια αργότερα να που συζητάμε για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής. Λέμε ότι θα εμπεριέχει και ένα μόνιμο σώμα με δύναμη 10.000 ατόμων. Συζητάμε επίση για τι νέε αρμοδιότητε του οργανισμού αυτού. Μα νομίζω ότι ο οργανισμό αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύη μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών, αν θέλετε, κρατών της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέκα άνθρωποι είναι στο κατάλογο για το CatchDI. Θα ήθελα πραγματικά να δώσω σε όλους το λόγο, όμως σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό που θα σας δώσουμε, διότι στις πέντε ψηφίζουμε και υπάρχει άλλο ένα θέμα στη διάταξη πριν. Οπότε σας ζητώ πολύ ευγενικά να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό της παρεμβάσης σας. Η κυρία Σρόιντοβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόταση σχετίζεται με το με πολύ μεγάλο λάθος που έγινε το 2015-2016 όταν τα εξωτερικά σύνορα της Σέγγεν δεν προστατεύθηκαν καταλήλως και υπήρξε διέλευση έως και 2 εκατομμυρίων ανθρώπων μεταναστών και προσφύγων. Κάποιοι από αυτούς ήταν όντως πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις φρικαλαιότητες του. Όμως πολλοί από αυτούς δεν ήταν επιλέξιμοι για άσυλο και θα πρέπει να επιστραφούν. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξωτερικά τη σύνορα για λόγους ασφαλείας. Όταν έχουμε εκατομμύρια ε, οι μετανάστες οι οποίοι περνούν τα σύνορα, τότε η αίσθηση για τι χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, μετά από τρία χρόνια ε, καλής λειτουργίας, η νέα αυτή υπηρεσία, λέει η κυρία Πίκουλα, ε, ο κύριο Πίκουλα θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντό της Σέγγεν. Καλωσορίζω λοιπόν την θέσπιση αυτής ε, της ε, ε, δύναμης είναι μια αντίδραση στους κινδύνους που υπάρχουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να εξετάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για την ε, χορήγηση ασύλου. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο Σέγγεν, έχει να κάνει και με την έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Είναι καλό ότι θα έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στίβενς, η κυρία Στίβενς. Κυρία, κυρία Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Πάντα είμαστε υπέρ του Frontex. Πρώτη φορά το 2016 ο Frontex ανέλαβε το καθήκον να παρεμβαίνει περισσότερο στις επιστροφές ε, μετά από απόρριψη ασύλου. Και τώρα ξανά υποστηρίζουμε τον Frontex. Γιατί πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Frontex έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. Μπορεί να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο με ισχυρά εξωτερικά σύνορα και εδώ θα μας βοηθήσει ο Frontex. Περισσότερο, περισσότερο πόροι, προσωπικό, θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα έτσι τις προκλήσεις. Ο Frontex θα πρέπει να δραστηριοποιείται και σε μη ε, κράτη-μέλη, ε, χώρες που βρίσκονται μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Frontex θα βοηθάει στις επιστροφές από το Μαρόκο προς μια άλλη χώρα μη μέλος, την Νιγηρία για παράδειγμα, τον Νίγηρα. Αυτό δεν μπορούσαμε, δεν το κάνουμε. Είχαμε χάσει αυτή τη δυνατότητα στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Να ε, πω ότι λυπάμαι ότι σε σημαντικό θέμα που ε, χιλιάδες ζωές εμπλέκονται και εκατομμύρια ε, ευρώ ε, δεν ε, γίνονται τακτές οι ερωτήσεις και δεν γίνεται καλή συζήτηση. Η λύση είναι το κράτος δικαίου. Αν, ο κόσμος, ε, ε, κάποιος επιδιώξει να μπει στην Ένωση παράνομα, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός κανόνας που θα λέει «Παρακαλώ, λυπάμαι, πρέπει να πάτε πίσω». Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει και νόμιμη οδός για την ε, αίτηση ασύλου γιατί όλα τα πολιτισμένα κράτη δέχονται το δικαίωμα του ασύλου για αυτούς που διώκονται. Το κράτος δικαίου είναι το βασικό. Τα 11 δις ευρώ και οι έξτρα πόροι και η γραφειοκρατία θα βοηθήσουν ε, ε, να λύσουμε το πρόβλημά μας, ε, ενώ ένας πρακτικός κανόνας θα ήταν καλύτερος. Μπόκοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να έχουμε ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στην Ευρώπη και προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο χώρος Σέγγεν. Δυστυχώς όμως δεν αντιμετωπίσαμε έτσι τα πράγματα του 2015. Επιτέλους όμως, τρία χρόνια μετά, συντοποιούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την παράτυπη μετανάστευση και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποια βήματα ακόμα. Η εντολή του Frontex θα πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, να μπορεί να περιλαμβάνει και τις επιστροφές από τρίτη χώρα προς τρίτη χώρα. Στη Σλοβενία το 2015 είχαμε σε καθημερινή βάση χιλιάδες διελεύσεις των συνόρων μας και είδαμε ότι η τάση είναι ανωδική και του τελευταίου μήνε. και δεν νομίζω ότι πρόκειται να τροποποιηθεί πολύ στο μέλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι έρχονται από τη Βοσνία ή τη Σερβία θα, μπορούν να, θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφονται χάρη στο Frontex. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι Ευρω... Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Ισπανός. Είναι πολύ καλή η στόχη ενό στόχου ε, ελευθερία ε, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ε, έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, και σε αυτό θα μας βοηθήσει η ακτοφυλακή, η συνοριοφυλακή ευρωπαϊκή με μια ε, νέα δυνατότητα 15.000 ε, ε, ανθρώπους με σημαντική χρηματοδότηση. Εμείς οι σοσιαλιστές ε, συνεισφέραμε στη βελτίωση του κειμένου με τροπολογίες για να μην υπάρξουν επιστροφές σε τρίτες χώρες και να το συνδέσουμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το των Θεμελιών Δικαιωμάτων που ισχύει. Όμως, πρέπει να ξέρετε ότι είναι αρκετά πικρό, πικρή η τελική γεύση, διότι υπάρχει τελικά μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και λιγότερη στον ανθρωπισμό. Στα νότια σύνορα της Ένωσης βρίσκεται η Ισπανία ε, και το πακέτο για το άσυλο ε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το, ο κανονισμό του Δουβλίνου επίση είναι μπλοκαρισμένο στο Συμβούλιο. Αυτά μένουν να γίνουν από το επόμενο Κοινοβούλιο. Ο κ. Μαριά έχει το λόγο, παρακαλώ. για άλλη μια φορά θέλω να μεταφέρω την κραυγή αγωνίας των κατοίκων των νησιών του αιγαίου για τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές και κυρίως το μεγάλο αριθμό παρανόμων μεταναστών οι οποίοι εισραίουν στην ελλάδα. πρόσφατα έγινε και εκδήλωση διαμαρτυρίας στην σάμο γιατί πλέον οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. πιστεύω ότι ο ρόλος της frontex πρέπει να βελτιωθεί να μπορέσει πραγματικά να κάνει σοβαρή δουλειά στα θέματα που αφορούν την φύλαξη των συνόρων όχι μόνο στα θαλάσσια σύνορα γιατί βλέπουμε πλέον μεγάλη έλευση και από την μεριά των χερσαίων συνόρων την περιοχή του εύρου. επομένως εδώ πρέπει να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη βελτίωση της δουλειάς που κάνει η ίδια η frontex αλλά και στην περιοχή της Υπήρου που υποτίθεται υπάρχει η frontex στα σύνορα ελλάδος αλβανίας και από εκεί έχουμε εισρωή κακοποιών οι οποίοι πραγματικά ληστεύουν τα παραμεθόρια χωριά. ευχαριστώ. Ο Σπισίλ, παρακαλώ.